διεξαγωγή ψηφοφορίας. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στα σοβαρά θέματα, δηλαδή στην διάταξη των εργασιών που έγινε δεκτή από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων ε, στη συνεδρίαση της 5ης 10 Σεπτεμβρίου με βάση το σχετικό άρθρο του κανονισμού και έχετε λάβει αυτή την διάταξη των εργασιών, το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Βλέπετε ότι το πρόγραμμα μας ε, είναι πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ακροάσεις ε, των επιτρόπων και θα ψηφίσουμε σήμερα για τις ε, εγκρίσεις